η συγγήτρια κυρία Φαν Νίδεν Χόιτζεν. Και παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν ήσυχα, ήσυχα και όχι ομαδών. Η κυρία Φαν Χόιζεν, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να ψηφίσουμε για σοβαρά νομοθετήματα. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Μια στιγμή. Με συγχωρείτε συνάδελφε. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι να δείξουμε αυρότητα και να αποχωρούμε με ησυχία από την αίθουσα. Αυτό ισχύει και για τους Προέδρους ομάδων, κυρία Χάμς, κύριε Φερχόφστατ. Bitte Κύριε witam państwa zapraszam do głosu sprawozdawcę panią Dyrmel Pantorotologu Stine Sigitri Kyria van Nuevenhuizen Dank wel voorzitter, commissaris Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να ψηφίσουμε για πολύ σημαντική νομοθεσία. Πρόκειται για την πρόταση αυτή που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις. Ξέρουμε ότι το τελευταίο καιρό έχουν γίνει διάφορες παρεπίσεις που έχουν τροποποιήσει την κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Ε, γίνονται παραπίσεις των δικτών όπως έγινε με το Λίμπορ και των δικτών αναφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών. Βέβαια υπήρξε πρόστιμο στην Deutsche Bank όσον αφορά το δίκτυο αναφοράς Libor. Η παραποίηση αυτή ισχύει για διάφορες ε, τράπεζες και πια έγινε σαφές ότι τέτοιου είδους παράνομες πράξεις πρέπει να είναι και ποινικά κολάσιμες. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς για να υπάρχει οικονομική σταθερότητα και να υπάρχει καλή ρύθμιση για να αποφεύγεται παραποίηση τέτοιων δικτών αναφορά στο μέλλον. Η νομοθεσία που θα ψηφίσουμε αύριο προσπαθεί να πετύχει τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος και να προστατεύσει την πραγματική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετές ρήτρε ασφάλεια για μεγάλου δείκτε αναφοράς όπω είναι το Λίμπορ ή άλλοι ε, δείκτες αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Όμως η ρύθμιση πρέπει να φροντίσει επίσης να καλύψει όσο γίνεται μεγαλύτερο εύρος τέτοιων δικτών, όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης ώστε να μπορούν οι επενδυτές να κρίνουν πού θέλουν να επενδύσουν και ανάλογα να πορεύονται. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν πολλές πληροφορίες και να υπάρχει όσο γίνεται μικρότερος κίνδυνος και να μην υπάρχει συγκέντρωση της αγοράς. Να έχει περισσότερη δύναμη στα χέρια του ο χρήστης, ο καταναλωτής τέτοιων δικτών και να υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα και στην οικονομία. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των δικτών αναφοράς απαιτεί καινοτομία, περιορισμό των κινδύνων και πειθαρχία στους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι για μικρότερους δείκτες αναφοράς πρέπει να υπάρχει διαφορετική ρύθμιση από ό,τι για τους πιο μεγάλους. Η έκθεση, έτσι όπως έχει σήμερα, προσπαθεί να πετύχει αυτή την ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών δικτών αναφοράς ε, μεταξύ εκείνων της αγοράς και των ε, προϊόντων, εκείνων που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Η ισορροπία αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία του καταναλωτή και για την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίου να υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες και ρυθμίσεις και οι σωστοί στόχοι ώστε να έχουμε μια νέα κατάσταση όσον αφορά την αγορά κεφαλαίων. Γι' αυτό ακριβώς με μεγάλη πλειοψηφία μόνο 10 κατά εγκρίθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και την στήριξαν και από τη δεξιά και από την αριστερά διάφορες πολιτικές ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεχητές, τον συνάδελφο Γιάλε, για παράδειγμα για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε προκειμένου να εκπονήσουμε την έκθεση αυτή. Προσβλέπω σε παρετέρω συνεργασία ώστε να προχωρήσουμε θετικά και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ζητάω από όλε τι πολιτικέ ομάδε να στηρίξουν την έκθεση αυτή ώστε γρήγορα και με μια ισχυρή εντολή να μπούμε σε τριμερή διάλογο. Έχουμε δύο χρόνια που συζητάμε, έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλή νομοθεσία για τους δείκτες αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νίουενχάουζεν. Ο Επίτροπος Χίλ τώρα. Παρακαλώ. Mr. President... Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι δείκτες αναφοράς ίσως φαίνονται ένα τεχνικό ζήτημα ίσονο σημασίας. Στην ουσία όμως σχετίζονται άμεσα με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία γενικότερα. Είναι η βάση κατάρτισης συμβάσεων. Ορίζουν την αξία χρηματικών προϊόντων καθώς και τα επιτόκια που καταβάλλονται στα ενυπόθηκα δάνεια και ε, τα, τις ε, συντάξεις για τον ορισμό των συντάξεων χρησιμοποιούμε επίσης αυτούς τους δείκτες αναφοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εμπιστευόμαστε τους δείκτες αναφοράς. Μία σειρά σκανδάλων όμως δυστυχώς έχει υποσκάψει αυτή την εμπιστοσύνη. Και μην ξεχνάμε ότι ε, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με χειραγώγηση το οποίο σημαίνει κλοπή και απάτη. Άρα για να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη θεωρούμε ότι οι πάροχοι δικτών αναφοράς θα πρέπει να την χάνουν ρύθμισης και εποπτείας. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, κυβερνητικοί έλεγχοι και να λύνονται θέματα που σχετίζονται με την διαφάνεια των δικτών αναφοράς και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα διασυνοριακής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει εποπτεία στα πλαίσια της ΕΣΜΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο θέμα, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο. Και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα στο τριμερή διάλογο να συζητήσουμε επιμέρους θύματα και πιστεύω ότι η εμβέλεια της νομοθετικής πράξης αφορά μικρούς και μεγάλους δείκτες αναφοράς. Γι' αυτό η ΕΚΟΝ έκρινε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση αποτίμησης κινδύνων όταν ορίζουμε τους δείκτες αναφοράς. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η πρώτη που θα νομοθετήσει επί του θέματος, θα πρέπει να ορίσουμε και το θέμα της πρόσβασης τρίτων χωρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, εισάγουμε κινδύνους. Θα πρέπει να έχουμε ένα εύρωστο σύστημα και να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Συνολικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα έτσι ώστε να οικοδομήσουμε ένα εύρωστο οικονομικό σύστημα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα ακολουθήσουμε και θα πρέπει να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Εξ της Επιτροπής Ήτρε, η κυρία Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η πλειοψηφία των πολιτών πλήττεται από αυτούς τους δείκτες. Έχουμε διάφορους ε, παρόχους που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες κατάρτισης δικτών. Έχουμε να κάνουμε και με δημόσια αγαθά, μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το εύρος της ζημίας της δημόσιας αγοράς λόγω της ε, χειραγώγησης των δικτών. Θα πρέπει λοιπόν να διώκονται όσοι παραποιούν τους δείκτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα βασικά προϊόντα ορίζονται από τους δείκτες αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ενέργειας. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ευαλωτότητα της αγοράς και της παραγωγής. Το εύρος των τιμών είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τους ε, ε, επενδυτές, αλλά και τον τελικό χρήστη, δηλαδή τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα ως προς την παροχή υπηρεσιών ενέργειας. Υπάρχει επίσης σύγκρουση συμφερόντων, γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Χαιρετίζω αυτή την ε, προσπάθεια και θα ήθελα να μειώσουμε την ευαλωτότητα και οι τιμές πραγματικά να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της αγοράς. Να έχουμε να κάνουμε με αξιόπιστους δείκτες έτσι ώστε να λευθούν δεσμευτικά μέτρα και κυρώσεις σε περίπτωση παραποίησης και χειραγώγησης η αποτίμησή μου είναι αρνητική. Όχι μόνο γιατί δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις μου, αλλά επειδή οι βασικοί δείκτες αναφοράς είναι πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες μας. Δεν υπάρχει αναλογικότητα και σωστός ορισμός ενός δείκτη αναφοράς συστημικής σημασίας. Οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι έχουν υποβάλει προτάσεις α, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πράξουμε και όχι να κάνουμε ότι πράττουμε. Θα πρέπει έτσι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά με πραγματικά μέτρα και επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο κύριος Νίντερμαγερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Κόρα Φανιούχαουζεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναγνωρίζουν το πρόβλημα όσον αφορά την αξιοπιστία των ε, αγορών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν αλευθεί διάφορα βήματα προκειμένου να υπάρξει ισορροπία και να γίνουν πιο γερές οι συναλλαγματικές ε, αγορές. Τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και έναν ε, πιο εύρωστο και ασφαλή χώρο. Πολύ καλά παρουσίασε την πρότασή της η συγγήτρια. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκε την προηγούμενη φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι βέβαια αρκετά τεχνική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει ότι είναι μια πρόταση σε βάθος που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που υπάρχουν για τους μικρούς δείκτες και ότι παραμένουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο είναι αρκετή η ρύθμιση αυτή στο σημερινό πλαίσιο βάσει των ε, ρυθμίσεων της Ιόσκο. Εγώ πάντως είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπόρεσα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια πάνω στην νομοθετική αυτή πρόταση. Επέλεξε μια ισορροπημένη πρόταση, ισορροπημένη ανάμεσα στη ρύθμιση των πιο σημαντικών ε, δικτών ε, αναφοράς, Αναφέρει όμως και τη διαφάνεια όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες. Πιστεύω ότι έτσι βελτιώνει την κατάσταση και όσον αφορά τις τρίτες χώρες και υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη των εθνικών ρυθμιστών και την ε, ευθύνη των υπολείπων. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ καλή πρόταση, πιστεύω. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας δώσει ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στον τριμερή διάλογο. ελπίζω να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατόν ρύθμιση, κάτι το οποίο όλοι βέβαια προσδοκούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα, Γιάννης Φερνάντες, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης εισηγητές που διαπραγματευτήκαμε πάνω στον κανονισμό αυτό τους τελευταίους μήνες. Πιστεύω ότι βελτιώνεται πάρα πολύ η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θέση της ομάδας μου, των σοσιαλιστών δηλαδή, ήταν ότι θέλουμε να βελτιώσουμε και να ρυθμίσουμε τους δείκτες με την πιο κρίσιμη σημασία. Σήμερα το πρωί καταφέραμε να καταλήξουμε και σε ένα αναπιωτικό ορισμό, ο οποίος να επιτρέπει να ορίσουμε και σε εθνικό επίπεδο τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας είναι δημόσιοι πολλές φορές όπως είπε και η συνάδελφος Ματίας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει μια λογική τιμή και ένας έλεγχος. Εξάλλου αυτοί οι δείκτες αναφοράς θα διέπονται από ειδικά σώματα όπως προτείνει και η ΕΣΜΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση στην οποία καταλήξαμε ώστε αυτοί οι δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, Λίμπορ κλπ. να διατηρούν την ισορροπία στην αγορά. Και οι δείκτες των πρώτων υλών επίσης να μπορούν να οριστούν ως κρίσιμη σημασίας. Η διαπραγμάτευση ήταν περίπλοκη. Χρειάστηκε να παραχωρήσουμε σε κάποια ζητήματα. Στο θέμα της αναλογικότητας αναφέρθηκε η συγκήτρια και άλλοι. Σημαίνει ότι οι μη κρίσιμη σημασία δείκτες θα ρυθμίζονται κάπως πιο περιοριστικά. Αλλά χάρη στην ομάδα μας, οι αρμόδιες αρχές της χώρας μέλη θα μπορούν να ελέγχουν και να εποπτεύουν τι κάνουν οι διαχειριστές με αυτούς τους δείκτες μη κρίσιμη σημασία. Να κάνουν δηλαδή ex μια ανάλυση των δικτών αυτών. Τέλος, καταλήξαμε σε συμφωνία προκειμένου οι δείκτες οι οποίοι καταρτίζονται σε τρίτες χωρές να καλύπτουν τους κανόνες της ΙΟΣΚΟ, κάτι το οποίο παλιά δεν ίσχυε. Είναι μια μεγάλη συμφωνία πάντως αυτή, η οποία θα επιτρέψει στους χρήστες, στους καταναλωτές να έχουν δείκτες πολύ πιο ικανοποιητικούς. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Τώρα, εκ μέρους του ECR, η κυρία Σουίμπερν. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ξεκινάω ευχαριστώντα την εισηγητρία για την πολύ σκληρή δουλειά τη. Υιοθέτησε μια λογική προσέγγιση και κατάφερε να ενώσει τόσε πολιτικέ ομάδε μια συμβαστική λύση που θα ψηφίσουμε αύριο. Πρόκειται για ένα πλαίσιο καλό, ώστε οι εθνικέ αρχέ να μπορούν να παρακολουθούν του δείκτε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι μπορούν και οι επενδυτές και οι καταναλωτές να την χάνουν προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά ορίζει ένα αυστηρό καθεστώς για τους κρίσιμη σημασία δείκτες χωρίς να επιβαρύνει ωστόσο ιδιαίτερα τους λοιπούς δείκτες. Ιδιαίτερη δίνεται έμφαση στην διαφάνεια για τον χρήστη και έτσι ο επενδυτής και καταναλωτής μπορεί να δηλώνει ο ίδιος αν ικανοποιημένο από την διαφάνεια και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δείκτης. Μια πιο ορθολογική λοιπόν προσέγγιση που ακολουθεί το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους μη κρίσιμη σημασία δείκτες είναι ευπρόσδεκτη. Αυτή όμως θα καταστεί δυνατή μόνο αν τα κράτη-μέλη καταστεί δυνατόν να υιοθετήσουν με ε, ορθολογικό τρόπο τους δείκτες οι οποίοι δεν θα μπαίνουν στην κατηγορία των κρίσιμου σημασίας δικτών ή αναλόγως αν θεωρούν ότι ένας δείκτης κινδυνεύει ε, να καταστρατηγηθεί να τον εντάσσουν στο εθνικό σύστημα των κρίσιμες σημασίες δικτών. Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να δώσουμε ε, προσοχή στις ε, τρίτες χώρες. Πρέπει οι αρχές της ΙΟΣΚΟ, της Εθνούς Ένωσης, να τηρηθούν και να βελτιώσουν έτσι τις προδιαγραφές βάσει των οποίων δρούν οι διαχειριστές των δικτών σε όλο τον κόσμο. Να μην γίνει δηλαδή αυτό που έχουμε δει με άλλα νομοθετήματα που είχαν και εκτός της Ένωσης εμβέλεια. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια καλή συνεργασία στον τριμερή διάλογο και να καταλήξουμε έτσι σε ένα κείμενο αποδεκτό και ικανοποιητικό για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σουίνμπερν, εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων, η κυρία Σιλβί Κουλάχ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστώ την ε, κόρα και είναι της ομάδας μου διότι όσοι ήταν από εδώ, εδώ από την προηγούμενη θητεία ξέρουν πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν το κείμενο που είχε να επεξεργαστεί και ελπίζω ότι τα λόγια αυτά που ακούστηκαν κύριε Επίτροπε όσο σκληρά και αν είναι θα σας καθοδηγήσουν στον τριμερή διάλογο ιδιαίτερα όταν θα έχετε να κάνετε με κράτη-μέλη τα οποία ίσως είναι υπερβολικά ε, διστακτικά ως προς την πρόοδο θα έχετε την δυνατότητα να εκφράσετε αντίστοιχα σαφείς διατυπώσεις και εναντί του. Το κείμενο λοιπόν της συναδέλφου για ορισμένα μου φαίνεται κάπως ασαφές ως προς το ρόλο της ΕΣΜΕ παραδείγμα της αρχής εποπτείας τραπεζών. Εγώ θα ήθελα να ήταν πολύ πιο σαφές ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να βγει εκτός παιδείας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να έχει βεβαίως το ρόλο που αναφέρει το κείμενο ε, στα τεχνικά ζητήματα, το τελικό διαιτητικό ρόλο για τον προσδιορισμό των δικτών κρίσιμη σημασία, που έχει πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως. Όλους αυτούς τους δείκτες που δεν έχουν νομισματικό ε, χαρακτήρα, χαρακτήρα δια τραπεζικών συναλλαγών ή ισοτιμίας, ισοτιμίας νομισματικής. οι δείκτες αναφοράς επίσης ε, θα είναι αρμοδιότητα τη ΕΣΜΑ. και νομίζω ότι όλες αυτές οι λύσεις είναι λογικές. Θα ήθελα και αν ήταν εδώ βέβαια το Συμβούλιο κύριε Πρόεδρε θα το επέκτηνα σε εκείνους ιδιαίτερα να επισημάνω το ζήτημα του προϋπολογισμού της ε, ΕΣΜΑ της Αρχής Εποπτείας ε, κινητών, της ε, Κινητών Αξιών και Αγορών που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να εξορροπηθεί και η πλαισίωση και υπό τη στενή έννοια εποπτεία τη της λειτουργίας ορισμένων δικτών και της αναλογικότητάς τους δεδομένου του μεγάλου αριθμού αυτών θα πρέπει να προχωρήσει βήμα το βήμα και ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να γίνουν και κάποιες μικροδιορθώσεις. Πάντως ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη για τον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Από την QNGL. Κύριος Χουάρης Θεαμπράντς, παρακαλώ, ένα λεπτό. Κύριε Χίλ, είπατε ότι όταν γίνεται παραποίηση αυτό σημαίνει απάτη, κλοπή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει ο στόχος να είναι η μείωση της παραποίησης των δικτών αναφοράς. Όμως ε, το νέο κανονιστικό πλαίσιο ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές είναι ανεπαρκές. Εάν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία για την ε, κατάρτιση του δίκτυ βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Βασιζόμαστε στην αρχή της ζήτησης και της προσφοράς. Θα πρέπει οι οικογένειες με λιγότερους οπόρους να μην πρέπει να ε, πληρώνουν περισσότερα ε, σε σχέση με τη χρήση του Eurobor ως προς το LIBOR. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγαλύτερη καταβολή. Ο κανονισμός αυτός δεν αφήνει περιθώρια ε, παρά την, ε, το γεγονός ότι οι τράπεζες δυστυχώς κάνουν πολλές υπερβολές και υπερβάσεις. Ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Αυτό που μας εκπλήσει με τους δείκτες αναφοράς είναι ότι οι παραβιάσεις κινούνται πέραν από την ε, οικονομική κρίση. Δυστυχώς, οι μεγάλες επιχειρήσεις, η Deutsche Bank και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυστυχώς παραπίσαν αυτούς τους δείκτες για δικά τους ε, κέρδη για πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί θα πούνε εντάξει σήμερα καταδικάστηκαν. Θα καταβάλουν χρηματικά πρόστιμα που θα πληρώσουν οι τράπεζες, όχι οι καταθέτες. Και σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει φορολογική ελάφρυνση όταν καταβάλλονται αυτές, αυτά τα χρηματικά ποσά, το οποίο σημαίνει ότι τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κόρα. Φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό μέχρι σχεδόν το τέλος. Στο τέλος όμως ορισμένες ε, τροπολογίες τελευταία στιγμής υποβάθμισαν τον κανονισμό, δηλαδή ε, αποσύρθηκαν ορισμένοι δείκτες κρίσιμης σημασίας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί δείκτες στην ουσία δεν εντάσσονται σε αυτή την νομοθεσία, γιατί υπάρχει άλλη διαχείριση των δικτών κρίσιμης σημασίας από τους κοινού δείκτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δέχτηκε μία πιο αυστηρή νομοθεσία όπως ε, ορίζουμε σήμερα, όπως είπε και η Σιλβί Γκουλάρ, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια ενιαία αγορά, τελικά επαφιέμεθα στα κράτη-μέλη χωρίς μεγάλο έλεγχο από την ΕΣΜΑ για, τον, ε, για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Άρα δεν μπορούμε να αφήσουμε να ορίσουν τα κράτη-μέλη τι είναι ένας δείκτης κρίσιμης σημασίας. Εάν αλλάξει αυτό το δεδομένο και την υπόψη της τροπολογίας μας, τότε θα υπερψηφίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από το EFTD, ο κύριος Γουλφ για ένα λεπτό. Δεν βλέπω εδώ τον κύριο Γουλφ. Ο κύριος Μονό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσέχοντας τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν για τους δείκτες αυτούς αναφοράς, καταλήγουμε να βρίσκουμε απογοητευτική την έκθεση αυτή με μια εποπτεία. Θα πρέπει πιο αυστηρά να ελέγχονται οι δείκτες αυτοί για να αποφεύγουμε τα σκάνδαλα του παρελθόντος. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και η δέσμευση αυτή έχει να κάνει μόνο με το u και το Libor. Θέλω επίσης να καταγγείλω και κάποιες ε, τράπεζες που είναι στην καρδιά των σκαδάλων και μας αναγκάζουν να δράσουμε. Το λίμπορ ήταν μια παραποίηση της αγοράς όπως έγιναν ε, και άλλες και προστίθεται στα διάφορα σκάνδαλα της HBCS και άλλων ε, φορολογικών πρακτικών, φοροαποφυγής δηλαδή κλπ. Η... Τα βάρη τελικά τα επομίζεται ο κόσμος. Αυτά τα οποία θα κερδίσουμε είναι ελάχιστα αν λάβουμε υπόψη μας τα εκατομμύρια κέρδη που βγάζουν αυτοί που κάνουν τις απάτες. Και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς να σπάσουμε αυτό τον ε, φαύλο κύκλο. Είναι προφανές ότι για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να υπάρχει έλεγχος στα εθνικά σύνορα των κεφαλαίων για να αποφεύγουμε την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ και τις ακάλυπτες πωλήσει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Παούνοβα έχει τώρα το λόγο. Τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εμπιστοσύνη στις αγορές μας επλήγει Εξαιτία τη παραποίηση δικτών αναφορά. Αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η εμπιστοσύνη πρέπει να ανακτηθεί. Το οικονομικό μα σύστημα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια. Γι' αυτό και χαίρομαι για την πρόταση αυτή και συγχαίρω όλου του συναδέλφου που δούλεψαν πάνω στην έκθεση αυτή γιατί δημιούργησαν έτσι ένα πλαίσιο για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Οι περισσότερες χώρες μέλη δεν έχουν κανόνες και κανονισμούς που αφορούν τους δείκτες αυτούς αναφοράς και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα αναρμονισμένο πλαίσιο για τους δείκτες αναφοράς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα οδηγήσει σε περισσότερη εμπιστοσύνη και σε καλύτερη και μεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα στην Ευρώπη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες των νέων κανόνων στην αγορά. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι μπορεί να δουλέψει πιο σκληρά, διαπιστώνει ότι μπορεί και να παρακάψει τους κανόνες. Αυτό όμως δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να μην βάζουμε επιπλέον βάρος πάνω στους διαχειριστές. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια με την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πέβανος Πεχές. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, Καταρχάς συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ τεχνικό αλλά και κρίσιμη σημασίας. Εν τέλει, συζητούμε το θέμα, το θέμα αυτό λόγω της Euribor και του σκανδάλου και λόγω του ζητήματος Libor. Διότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, να παρεμποδίσουν τη λειτουργία τους και τελικά να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτό χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθεί. Εδώ βρισκόμαστε ενώπιον μιας συμβιβαστική λύσης. Λυπούμε που οι εξουσίε της αρχής εποπτείας, αρχής η οποία δείχνει καθημερινά και αποδεικνύει την νυφαλιότητα των αναλύσεων και συστάσεών της δεν ενισχύονται ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον προσδιορισμό των κρίσιμων δικτών και την εποπτεία αυτών. Ιδιαίτερα δεν λυπούμε, διότι αφήνεται πολύ μεγάλο περιθώριο διακριτικό στα κράτη ως προς τους μη κρίσιμη σημασίας δείκτες. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μια απαιτητική νομοθεσία θα εξετάσει δε και την ε, ε, ισοδυναμία της με νομοθεσίες σε άλλες περιοχές του κόσμου επί τη βάση των υφισταμένων ε, διατάξεων ανεξαρτήτως των όσων γίνονται εδώ και μέσα στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Ένωσης νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αλλά πάντως εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στην πραγματευτική μας ομάδα Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας Δείχνω ανοχή, αλλά και η ανοχή έχει τα ωριά της. Ο κύριος Όζοκ έχει το λόγο τώρα. ECR, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση έχει πολύ σοβαρές και εύστοχες λύσεις για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις. Ευπρόσδεκτη λοιπόν η πρωτοβουλία, ευπρόσδεκτη η λύση για τους κρίσιμες και μη κρίσιμης σημασίας δείκτες. Επίσης συμφωνώ στα όσα λέγονται για την ΆΙΟΣΚΟ, για τη Διεθνή Ένωση και για τους ε, δείκτες και δείκτες που εφαρμόζουν τρίτες χώρες. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε τους κανόνες αυτούς, οι δείκτες θα λειτουργούν πιο ομαλά, θα είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε χειραγώγηση και άρα θα ανακτήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη για τις χρηματοποιητικές ε, αγορές. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια στις διατάξεις τις σχετικές με το πεδίο εφαρμογής και καταλληλότερη νομοθεσία ως προς τις παρεκκλήσεις για ορισμένες κατηγορίες διαχειριστών. Ε, Επίση, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, η σαφήνεια καλύτερα για του μεταβατικούς κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Πάτρικ Οφλίν. Δεν εδώ κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε Χίλ εύρωστοι και διαφανείς δείκτες είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς, για μεγάλων αξιών ε, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις που εξαρτώνται από τους δείκτες και έχουμε ιδιαίτερα δώσει έμφαση όλοι στην αρχή της διαφάνειας. Ήδη αναφέρθηκε το σκανδαλό Λίμπορ νωρίτερα. Αποδεικνύεται ότι η διαφάνεια είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση συμφερόντων και οι καταστρατηγήσεις, οι χειραγωγήσεις. Κατέστη σαφές από το σκάνδαλο Λίμπερ ότι εάν δεν υπάρχει διαφάνεια δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόθεση χειραγώγησης από τους διαχειριστές, όπως είδαμε με την Deutsche Bank και το σκάνδαλο Λίμπορ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και οι διαχειριστές να ε, παρακολουθούνται στενά θα πρέπει επίσης ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουμε ρύθμιση για καλύτερη μακροοικονομική ε, εποπτεία. Αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα για την απρόσκοπτη λειτουργία του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα, κυρία Κάπελ. No. Okay, uh, please take Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω τη κυρία Κάπελ να τη ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, οι παραπίσεις που έλαβαν χώρα στις αγορές, πολλές από αυτές έγιναν από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από μεγάλες τράπεζες. Και τελικά τους κρίσιμες σημασίας δείκτες αφήνουμε να τους καταρτίζουν μανωμένα διάφορες χώρες. Δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να επιβάλλει για τους κρίσιμες σημασίας δείκτες να επιβάλλονται οι κανόνες εξίσου σε όλες τις χώρες μέλη και σε όλα τα χρηματοπαιδευτικά ιδρύματα. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ήταν η ερώτηση του κύριου Φρουνσούλητσα, παρακαλώ. Νομίζω ότι η πρόταση είναι πολύ ε, ε, καλό μείγμα, ε, ισορροπημένο μείγμα λύσεων για τους κρίσιμης σημασίας δείκτες, για πρώτες ύλες κτλ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η έκθεση λύνει με αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο τα προβλήματα ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το σημείο εκκίνησης είναι εξαιρετική εργασία για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, διότι τηρεί τον απότερο στόχο μας. Με βάση την κρίσιμη κατάσταση που ισχύει, θα πρέπει να οικοδομηθεί εκ νέου ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Τα σκάνδαλα είναι καταδικαστέα, αλλά δεν θα πρέπει να προωθήσουμε και έναν ψυχολογικό πόλεμο. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι έφτασε σε μία σωστή εξισορρόπηση. Είδε ποιες είναι οι διακρίσεις μεταξύ δικτών κρίσιμης σημασίας και δικτών που δεν θεωρούνται χρήσιμοι και στη χώρα μου στην Ιταλία αντιμετωπίσαμε μία ε, δυσκολία σε σχέση με τους κινδύνους και τις ζημίες που υπέστησαν 2,5 ε, εκατομμύρια νοικοκυριά. Και λέμε και συζητάμε το γεγονός ότι η Deutsche Bank προώθησε παράγωγα που είναι πέντε φορές το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λύσουμε το πρόβλημα, όχι να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση τρόμου. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Σαλίνη. Πώς πιστεύει ότι θα εκδηλωθούν οι συνέπειες αυτών των μέτρων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορεί να εξελιχθεί η γραφειοκρατία στον τομέα αυτόν ώστε να έχουμε στο δυνατόν πιο θετικές εξελίξεις. Ευχαρίστως να απαντήσω στον κύριο Ρούμπιχ οι ανησυχίες μας ε, σε σχέση με τις επιπτώσεις της ΜΜΕ είναι μια ανησυχία που συμμερίζομαι και πολλές φορές ε, απαντώ με δυσκολία γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, επιπτώσεις που δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων ο δρόμος είναι ο σωστός και θα πρέπει να επιβάλλουμε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να θέσουν στο κέντρο των μελημάτων τους της ΜΜΕ. Αυτό σημαίνει και αναθεώρηση της διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όχι μόνο να ορίσουμε τους δείκτες αναφοράς. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω την ε, κυρία Νίνα Τζιλ. Οπότε ο κύριος που έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι η παραποίηση του Λίμπορ και άλλων δικτών που έγιναν από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέληξε σε καταστάσεις όπου επιχειρήσεις και επενδυτές έχασαν πάρα πολλά χρήματα. Οι ρυθμιστές των οικονομικών αγορών αποφάσισαν να επιβάλλουν κυρώσεις. Κυρώσεις εκατομμυρίων ε, ευρώ. Όμως αν συγκριθούν με τις απώλειες των επενδυτών Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τώρα μέτρα τα οποία να μας βοηθήσουν πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τέτοια σκάνδαλα στο μέλλον. Η έκθεση αυτή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει τρεις στόχους. Πρώτον, να τεθούν οι προδιαγραφές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους κρίσιμες σημασίες δείκτες αναφοράς και επίσης θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνονται τέτοιες ε, παραπίσεις. Δεύτερον, μεγαλύτερη διαφάνεια, να υπάρχει πληροφορία και ενημέρωση για όλους τους χρήστες, για όλους τους δείκτες αναφοράς, να είναι καλά ενημερωμένοι πριν πάρουν την όποια απόφασή τους και τρίτον να υπάρχει πρόσβαση για την διαχείριση των ε, δικτών αυτών αναφοράς. Ελπίζω όταν θα εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή μάλλον θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε να μην υπάρχουν τέτοια σκάνδαλα, να μην εμφανιστούν τέτοια σκάνδαλα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν έτσι συνεκτικός. Ο κ. Μπούντα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κεντρικό μέλημα την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Υπ' αυτή την έννοια τα χρηματοοικονομικά δοτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για, τη, για τις συμβάσεις θα πρέπει να διέπονται από μια διαφανή νομοθεσία. Συνεπώς, ε, κατανοούμε ότι οι δείκτες αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ε, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε στρέβλωση των πραγματικών καταστάσεων. Θα πρέπει να ορίσουμε υπεύθυνου ε, φορείς και μέσα έτσι ώστε να αποθαρρύνουμε τις παραποίησεις. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλές φορές οι αγορές διαφέρουν από την πραγματική οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δείκτες αναφοράς, αφήνοντας όμως ε, τους μηχανισμούς αυτούς στα εθνικά κράτη-μέλη. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προδιαγραφές των συστημάτων διακυβέρνησης για να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Μόνο τότε θα υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, ίσως ανταγωνισμός και όχι αθέμητος, ούτε έναντι τριών, τρίτων χωρών. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζει η διαδικασία Catch the Eye. Μαριάννα Πέτια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή θέλει να προσφέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για τις διάφορες ε, συμβάσεις. Ο κύριος στόχος είναι η προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλους τους δείκτες αναφοράς που καθορίζουν την ε, τιμή, την αξία μιας σύμβασης ενός συμβολέου ή καθορίζουν ε, την καλή απόδοση. Η ακρίβεια, η εγκυρότητα των δικτών είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για την έκθεση αυτή. Στηρίζω λοιπόν τους κύριους στόχους που είναι η βελτίωση του πλαισίου που καθορίζει τους δείκτες αναφοράς. Οι επιπτώσεις οι δημοσιονομικές δεν πρέπει να μας εμποδίσουν να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι το πλεονέκτημα μιας καλής διαχείρισης των δικτών αναφοράς, κρίσιμης σημασίας και ο έλεγχος εκείνων που δεν είναι κρίσιμης σημασίας αξίζουν τον κόπο. Η περίπτωση παραποίησης των δικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και οι παραποίησεις που έγιναν στον τομέα της ενέργειας μας δείχνουν ότι έχουμε την υποχρέωση να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Νικόλα Καπούτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να τύχουν χειραγώγησης με βάση τους δείκτες αναφοράς για τη χειραγώγηση του ΛΑΙΜΠΟΡ και του EURIBOR. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ευαλωτότητα της αγοράς για να μην υπάρξουν ζημίες κατά των καταναλωτών και των τελικών χρηστών. Γι' αυτό θα πρέπει να επανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών ορίζοντας στους δείκτες αναφοράς. Συμφωνώ λοιπόν ε, με την έκθεση ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέσα σωστής διακυβέρνησης για να, αρθούν και, να αρθεί και η σύγκρουση συμφερόντων ορίζοντας ε, εξισορροπημένες αρχές διακυβέρνησης έτσι ώστε να έχουμε σωστούς δείκτες αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες κρίσιμης σημασίας ή συστημικούς δείκτες γιατί δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την χειραγώγηση των δικτών από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, γνωστή τραπεζική κολοσσή όπως η Deutsche Bank τιμωρήθηκαν με πρόστιμα γιατί χειραγώγησαν τον δίκτυο αναφοράς Libor, κερδίζοντας έτσι παράνομα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ όμω αυτό δεν φτάνει αφού μετά την οικονομική κρίση οι τράπεζε που διασώθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων ασκούν τη σκληρή και ανάλγητη πολιτική του ενάντια στους μικροδανειολήπτε και βγάζουν στο σφυρί χιλιάδε σπίτια στη Νότια ευρώπη. μεγάλο πρόβλημα στην ελλάδα έχει επίση δημιουργηθεί για του μικροδανειολήπτε στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο έτσι πάνω από εβδομήντα χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν σε δυσχερέστατη θέση όσον αφορά το κόστος αποπληρωμής των δανείων τους μετά τη σοβαρή μετατροπή ισοτιμίας ευρώ ελβετικού φράγκου αφού οι τράπεζες κατά παράβαση του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης για τους καταναλωτές δεν τους ενημέρωσαν ότι κάθε καταβαλλόμενη μηνιαία δόση επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής. πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των δαλειοληπτών στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο που μόνο το τελευταίο διάστημα λόγω της μεγάλης πτώσης του ευρώ έχουν χάσει επιπλέον πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι στηρίζω την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι η συγγήτρια πολύ σωστά την έχει ετοιμάσει. Έτσι σταματάνε οι δυνατότητες παραποίησης από πλευρά των τραπεζών και σταματούν και τα σκάνδαλα που διαπιστώσαμε τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Πρέπει να ενισχύσουμε τη σταθερότητα του δημοσιονομικού μας συστήματος και πρέπει να έχουμε μια καλή αγορά κεφαλαίων. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στις αδικίες και η απάτη που έχει να κάνει με την, ε, το ελβετικό φράγκο όπου οι τράπεζες γέμισαν τις τσέπες τους ενώ οι πολίτες εξαρτώνται τώρα από τα δάνειά τους και κινδυνεύουν. Όντως αξίζουν την αλληλεγγύη μας. Ως πολιτικοί πρέπει σε τέτοιους χώρους να τα λέμε αυτά. Γιατί τέτοιες συζητήσεις παρακολουθούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριος Γλέζος. Αδελφοί, το σκάνδαλο με τη Deutsche Bank μου θυμίζει το, ε, τον επέσχυντο ρόλο που έπαιξε η Deutsche Bank στη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα όπου ξεζούμισε κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό και επειδή ακόμα η Γερμανία δεν εκπληρώνει τις οφειλές προς την Ελλάδα η Deutsche Bank συνεχίζει το καταστρεπτικό ρόλο. Το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι μήπως ματαιοπονούμε για τη σωτηρία των τραπεζών με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο όπου ό,τι έγινε στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα χρόνια ξεζούμισαν τον ελληνικό λαό για να σωθούν το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. αναφέρω ένα συγκεκριμένο γεγονός η τράπεζα της ελλάδος αποκάλυψε ότι από το 2010 έως το 2014 πήραμε 226 δισεκατομμύρια ευρώ και δώσαμε 270 δισεκατομμύρια ευρώ. 33 δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτό και μόνο προσδιορίζει το επέσχυντο όλων των προσπαθειών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίγκορ Σόλτερς. Πρόεδρε. Μπορούμε να πούμε επιτέλους πια κατατέθηκε η πρόταση. Ο καρονισμός μπαίνει προς την ορθή κατεύθυνση. Γιατί από τους δείκτες εξαρτώνται πολλά χρηματοπιστωτικά εργαλεία ύψους ε, πολλών εκατομμυρίων και αντίστοιχα επενδύσεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων και ενυπόθηκα δάνεια. Οπότε η καταστρατήγηση αυτών των δικτών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικές απώλειες για τον καταναλωτή και τον επενδυτή. Πρέπει να είναι σταθερή η αγορά. Έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια πολλή κερδοσκοπία, πολλές χειραγωγήσεις. Έχουν μετατραπεί αυτές σε εργαλείο για την δημιουργία πλασματικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, το οποίο διοικεί ολόκληρο τον κόσμο πλέον. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και να προβλέψουμε κυρώσεις και μηχανισμούς εποπτείας. Σας ευχαριστώ πολύ και εν τέλει Ο κύριος ε, much. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε το γεγονός ότι στην έκθεση αυτή η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, εξασφάλισε μια ε, υγεία οσορροπία μεταξύ κρίσιμων και μη δικτών και αυτών που αφορούν τα βασικά αγαθά. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, και λοιπόν, αντίκειμε απολύτως στην ιδέα του προσδιορισμού των κρίσιμης σημασίας δικτών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει την αποτροπή σκανδάλων και καταστρατηγήσεων της αγοράς που είδαμε στο παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές για μια καλή και ισορροπημένη πρόταση που είδαμε εν τέλει στο κείμενο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Χιλ. Έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τις κυρίες και κύριους βουλευτές για τις τοποθετήσεις τους. Ήταν εξαίρετη η συζήτηση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σημειώσω ότι επικρατεί ευρύτατη συμφωνία. Συμφωνία ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να θέσουμε ένα τέρμα στις χειραγωγήσεις που έχουμε δει να εκδηλώνονται τόσο συχνά στο παρελθόν. Συμφωνία ότι είναι πολύ σημαντική η αρχή της διαφάνειας ότι είναι πολύ σημαντική η καλύτερη διακυβέρνηση, συμφωνία ως προς την ανάγκη για καλύτερη νομοθεσία και εποπτεία. Ε, συμφωνούμε λοιπόν ότι έχει εξασφαλίσει ένα πολύ καλό πλαίσιο η συγγετρία και έτσι αντιλαμβάνουμε ότι ορισμένοι θα ήθελαν πιο αυστηρές διατάξεις ως προς την εποπτεία ή ως προς τον ορισμό των μη ε, κρίσιμης σημασίας δικτών εν τέλει. Αλλά έχοντας ακούσει τη συζήτηση είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί το κατάλληλο κοινό έδαφο ώστε να προχωρήσουμε ταχύτατα στην υπόθεση αυτή προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος των επενδυτών, προ όφελο της εμπιστοσύνης της αγοράς και εν τέλει προς όφελος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Χρειαζόμαστε τις ε, διασφαλιστικές αυτές τις δικλείδες το ταχύτερο δυνατό. Πολλοί από τους ομιλητές επεσήμαναν ότι χρειάστηκε να περάσει πολλής χρόνος για να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε αυτήν την πρόταση και να την ε, σπρώξουμε με ούριο τον άνεμο όπως νομίζω φαίνεται να έχουμε. Θα δώσουμε μεγάλη όθηση λοιπόν έτσι στις χρηματικές αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτρέψουμε καταστρατηγήσεις και θα αποτρέψουμε εσφαλμένη περιγραφή κρίσιμης σημασία δικτών. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια και τους κοιότητες εισηγητές για την πολύ σκληρή δουλειά τους. Ήταν κρίσιμη και αυτή η κρίσιμη σημασία για την πρόθεση του, της προτάσεως και πιστεύω ότι θα έχουμε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο για να καταλήξουμε ταχύτητα σε ένα νομοθέτημα, σε ένα τομέα που πρέπει ταχύτατα να ρυθμιστεί νομοθετικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η συγκεκριά μας τώρα, η κυρία Κόρα Φαν Νιουβενχόιζεν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους, για τις τόσο αξιόλογες παρατηρήσεις τους και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τη στήριξή τους. Φυσικά δεν είναι ικανοποιημένοι όλοι 100% αλλά η έκθεση στο σύνολό της νομίζω ότι αξιολογείται θετικά. Δέχομαι ευχαρίστω στα συγχαρητήρια, αλλά θέλω να τα μοιραστώ με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, με βοήθησαν πάρα πολύ και την πέτρα από την ε, συμβουλευτική πολιτική, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Ήταν η πρώτη μου έκθεση και ήταν ε, πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια που έκανα για να τηρήσω όλες τις διαδικασίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε χαίρομαι πολύ που τα κατάφερα. Και στον κύριο Μονό θέλω να πω ότι Οι κρίσιμη σημασία ε, δείκτε δεν είναι μόνο Libor και Eurobor, είναι και άλλοι. Συμφωνώ ότι εκτός από τα ποσοτικά κριτήρια πρέπει να υπάρχουν και τα ποιοτικά κριτήρια και αυτό έχω πει και εγώ ότι πρέπει να γίνει, γιατί μόνο έτσι θα ξέρουμε αν κάποιο δείκτη αναφοράς είναι κρίσιμη σημασία ή όχι. Δεν εξαρτάται μόνο από το κόστο του. Ευχαριστώ πολύ πάντως όλους και προβλέπω και εγώ σε καλή συνεργασία με τους σκιώδες εισηγητές και την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον τριμερή διάλογο. Να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή ρύθμιση για τους δείκτες αναφοράς. ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, πρώτη σας φορά. Συγχαρητήρια ακόμα περισσότερο. Πολύ καλά τα καταφέρατε.